Ε, που ξέρουν ακριβώς ε, ότι χρησιμοποιούν την πνευματική διοίκηση άλλων και κερδίζουν πολλά χρήματα στοχεύουμε ακριβώς σε αυτές. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα εφαρμοστεί τεχνικά το μέτρο αυτό που οι πλατφόρμες καλούν ε, τους χρήστες να αναφορτώσουν ό,τι επιθυμούν ακριβώς. Θα, θα πρέπει όμως να υπάρχει ευθύνη για τις ε, πλατφόρμες. Θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη σωστής ε, χρήσης των δικαιωμάτων μας και ιδιοκτησίας άλλων ή τη πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Νομίζω ότι με τη δουλειά που κάναμε έχουμε μια πολύ καλή βάση, ε, βάση ε, τη οποία μπορούν πλέον να δώσουν ε, τι οδηγίε του στα κρατημέλη για το πώ θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η οδηγία σε κάθε κράτο. Αυτό νομίζω ότι ήταν ο σωστό δρόμο, είναι ο σωστό δρόμο για να προχωρήσουμε προ τα επόμενα και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ελευθερία έκπραση, ψηφιακού κόσμου και πνευματική ιδιοκτησία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, τον κύριο Ντάντι. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Οπωσδήποτε χρειάζεται αναθεώρηση του κοινοτικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα. Η οδηγία καταδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο πολλές φορές δέχτηκε αυτή την αρχή, ιδιαίτερα ως προς την εξισορρόπηση των πλατφορμών. Ο βομβαρδισμός ε, στην ψηφιακή αγορά δείχνει ότι προσπαθεί κανείς να ξεφύγει από το πραγματικό περιεχόμενο. Δεν είμαστε υπέρ της λογοκρισίας. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει διάδοση πληροφοριών σε σχέση με κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ως προς τις ψευδείς ειδήσει υπάρχουν αυτοί που θα ήθελαν το δίκτυο να είναι μια άγρια δύση των μεγάλων πλατφορμών. Όμως θέλουμε να ανταμείψουμε του, τα πνευματικά δικαιώματα και τους δημιουργούς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Η Επίτροπος Γκάμπριελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητή, αγαπητέ εισηγητά, σκιώδης. Θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Η οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ψηφιακής αγοράς, της ενιαίας μας αγοράς αναγνωρίζουμε ότι μία προσωρινή πολιτική συμφωνία εξευρέθη για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Αγαπητά μέλη, πρόκειται για ένα ε, σημείο ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή πνευματική κληρονομιά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Η νέα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα μας επιτρέπει να φτάσουμε στους κοινούς στόχους σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα του 21ου αιώνα η οδηγία τάσεται υπέρ εκείνων που προασπίζονται, που προασπίζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Πρόκειται για τους εκδότες, παραγωγούς έργων, τις ψηφιακές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, συγγραφείς και ούτω καθεξής. Υπερασπίζεται τη δημιουργία και την τεχνητή ευφυΐα έτσι ώστε η πνευματική μας κληρονομιά να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες. Για πρώτη φορά στην νομοθεσία μας η μεμονωμένη πνευματικοί δημιουργή θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους θέση και θα μπορούν να έχουν μία σωστή ανταμοιβή. Αγαπητά μέλη, όλοι αυτοί οι δημιουργοί αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η πολιτιστική μας ε, κληρονομιά και η δημοκρατία μας. Αυτό ζητούν οι δημιουργοί. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι εξισορροπημένο αλλά και φιλόδοξο έτσι ώστε οι δημιουργοί και όσοι κατέχουν πνευματικά δικαιώματα να μπορέσουν να ανταμείβονται σωστά. Οι πάροχοι υπηρεσιών επίσης θα ανταμείβονται όπως πρέπει, καθώς και η δημιουργοί γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε μία ανακοίνωση για την ε, ε, κατάσταση σε σχέση με την ε, μετάδοση αθλητικών γεγονότων και το κείμενο προσαρτάται στο ε, στην οδηγία νομοθετικού περιεχομένου, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αναμένω τις ε, δικές σας, τη δική σας γνώμη και πιστεύω ότι με την υποστήριξη της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα θα αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα υπέρ των δημιουργών μας και των εν γέννη αξιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Για ένα λεπτό, ο κύριος Κρασμετόρσκι από την Επιτροπή ΙΤΡΕΜ. Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία είναι απαραίτητη. Το γνωρίζουμε όλοι. Όταν οι οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκαν πριν από καιρό, Νομίζαμε ότι θα ίσχυαν για πολύ καιρό και όμω ε, ήδη είναι πεπαλαιωμένε. Μάλιστα σε ορισμένε περιπτώσεις διαβρώνουν, διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Νομίζουμε ότι τα είχαμε κάνει όλα και όμως όχι. Το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα. Το διαδίκτυο είναι πεδίο μάχης για τους κολοσσούς της πληροφορίας με αποτέλεσμα να πιέζονται, να στριμώχνονται στη γωνία δημιουργοί και ερμηνευτέ. Οι οποίοι εν τέλει δεν αμείβονται για το έργο τους. για να μην πω ότι είναι θύματα εκβιασμού. Επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι μουσείων, δημιουργοί, περιμένουν λύση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναβάλουμε την απόφαση για την επόμενη ολομέλεια. Δεν είμαστε ακόμη όριμοι να πάρουμε απόφαση. Από την πολη Ζουλό. Κυρία Πρόεδρε, τα πλεονεκτήματα τα ανέφεραν άλλοι. Δεν θα τα επαναλάβω. Το ερώτημα είναι ένα. Τι σημαίνει αυτή η ψηφοφορία για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει τη χαρά να είναι μπροστά στην ψηφιακή ρύθμιση και να αποτελεί υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλουμε πλειοψηφία είτε για να συνεχίσουμε να είμαστε στο προσκήνιο πρωτοπόροι είτε για το αντίθετο. Η ψηφορία αφορά δυστυχώς το όλα ή τίποτα. Το θέμα είναι εάν ε, θα υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των μεν ή των δε. Εμείς θέλουμε να ωφελήσουμε τους πολίτες, τους δημιουργούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κόσμος θέλει ένα δίκαιο διαδίκτυο με ανοιχτέ πλατφόρμες όπου αμείβονται οι δημιουργοί και οι ερμηνευτέ, όπου προστατεύονται τα δικαιώματα. Αυτό ακριβώς λέει το κείμενο το οποίο ψηφίζουμε και η ψηφοφορία μας αφορά ένα θέμα οι πλατφόρμες έχουν ή όχι ευθύνη έναντι της κοινωνίας μας. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα στο οποίο καλούμεθα να απαντήσουμε. Και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη είναι υπέρ ενός ναι. Και λεπτό, Μπονή, Το άρθρο 13 σε διάφορε αμφιβολίε από την αρχή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και και χρειαζόμαστε μια συμβαστική λύση. Το διαδίκτυο δεν είναι απλώ η πρόσβαση σε διάσημου δημοσιογράφου. Είναι χώρο δημιουργία, ψηφιακή δημιουργία μάλιστα, και το χρησιμοποιούμε όλοι. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθηση. Πρέπει να ελέγχουμε και να ελέγχουμε και τα δικαιώματα. Εάν εσείς προωθείτε το προϊόν σας, το παστή ενδεχομένω, γιατί όχι. Και αυτό το αναγνωρίζει η μηχανή, το φίλτρο, οι πλατφόρμες. Και εκεί οι πλατφόρμες θα είναι προσεκτικές. Και ως προς το περιεχόμενο, ούτως ή άλλως αποφασίζετε εσείς. Στο παρελθόν, υπήρχε η γνωστή σε όλους μα λογοκρισία. Σήμερα όμως αυτό είναι λάθος. Είμαι υπέρ της διαγραφής του 13 και τότε και μόνο τότε θα υπερψηφίσω μια κατά τα άλλα πολύ καλή οδηγία. Και συγχαρητήρια στον Άξελ με την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Συναδελφοί, ε, σας άφησα λίγο περισσότερο χρόνο για τους εκπροσώπους των επιτροπών θα είμαι πιο αυστηρή μας από εδώ και πέρα. ποντά. ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεταρρύθμιση του τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων για τους χρήστες, τον, για τις πλατφόρμες, για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Και χαίρομαι που η πρόταση αυτή, η οδηγία αυτή, προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών και την πολιτιστική κληρονομιά. Χαίρομαι που προστατεύονται έτσι τα δικαιώματα όσων δημοσιεύουν και κάνουμε και κάτι για τις πλατφόρμες που παρανόμως διαδίδουν περιεχόμενο. Δεν πρόκειται προφανώς για λογοκρισία. Η λογοκρισία στο διαδίκτυο θα ήταν κάτι διαφορετικό. Θα, ήταν... είχαμε λογοκρισία αν αποτρέπαμε δημιουργούς, δημιουργικούς ανθρώπους να κερδίσουν αξιοποιώντας το ταλέντο τους στο διαδίκτυο. Δεν θέλουμε να τους ε, στείλουμε στην παρανομία ή σε μερική επασχόληση αφού πέρασουν μια μέρα οδηγώντας ταξί. Λοιπόν, χαίρομαι για το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Ήταν καλύτερο από ό,τι ανέμενα. Η κυρία Γκέριγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια συζητήσαμε διάφορες εκδόσεις του άρθρου 13 και τώρα καθίσταται σαφές ότι αυτό το κείμενο θα αλλάξει το διαδίκτυο όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα και θα υπάρχουν πολύ αρνητικοί αντίκτυποι στον ε, επιμερισμό της γνώσης. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς, αλλά στο τέλος τέλος ε, δεν φτάνουμε σε μια σωστή εξισορρόπηση. Είναι μεγάλο σφάλμα. Άρα η μόνη μας επιλογή είναι να διαγράψουμε το άρθρο 13. Αυτός είναι απαράβατος όρος έτσι ώστε οι ψηφιακές επιχειρήσεις να μπορέσουν να δράσουν γιατί ήδη έχουν αντιδράσει σε αυτό το κείμενο. Η εντολή που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να υπερασπιστούμε τις ΜΜΕ από το άρθρο 13 Δυστυχώς όμως θα είναι αναγκασμένες να αγοράσουν ε, ακριβή τεχνολογία φιλτραρίσματος που διαθέτουν μόνο οι Αμερικανοί γίγαντες. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουν προσπάθειες για, οποιαδήποτε, ε, για οποιοδήποτε πλαίσιο αδειοδότησης. Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ρόντε. Κύριε Ρόντε, ίσως μπορείτε να ασχοληθείτε με το θέμα κατά το χρόνο μιλία σας. Ο κύριος Καρίμ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Άξελ για αυτή την εξαιρετική εργασία. Συνάδελφοι, η δική μου προτεραιότητα είναι να καταστήσω σαφές ότι οι δημιουργοί θα μπορούν να ζήσουν στα πλαίσια της άσκησης των δικαιωμάτων τους, ε, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας με το κοινό. Αυτό είναι αναγκαίο με βάση τα νέα μοντέλα και πλατφόρμες που υπάρχουν. Δεν ήταν εύκολη διαπραγμάτευση, αλλά είμαι ικανοποιημένος γιατί φτάσαμε στους στόχους και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Γι' αυτό θα υποστηρίξω την έκθεση κατά την ψηφοφορία γιατί έχουν πολλές βελτιώσεις. Η εξόριξη δεδομένων θα είναι δυνατή για εμπορικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά. Το άρθρο 11 βελτιώθηκε έτσι ώστε η βιομηχανία δημοσιεύσεων να είναι ασφαλής. Θα μιλάμε μόνο για μικρές εξορίξεις οι οποίες εξαιρούνται επιγραμμικά. Επίσης, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εμπόρευσης των δεδομένων μέσα στα πλαίσια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Και συνεχίζεται ο κατάλογος. Υπάρχει ευελιξία για τα κράτη-μέλη και δεν θα υπάρξει εποπτεία των χρηστών. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες πλατφόρμες προσπαθούν να πείσουν διαφορετικά το κοινό, στην ουσία το κοινοβούλιο ε, δεν θα δεχτεί αυτή τη ροπή πραγμάτων που προωθούν ορισμένες πλατφόρμες. Κύριε Ρόντε, διαδικαστικό. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Είναι παράλογο ότι αποτρέπεται τη δεξαγωγή συζήτηση. Μας βλέπει σήμερα όλος ο κόσμος. Και έρχονται όλοι εδώ, στην Ολομέλεια, για να διαβάσουν τον λόγο που φτιάξαν στο σπίτι τους, αλλά συζήτηση δεν έχουμε. Αλλά το θέμα παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εσείς αποτρέπετε αυτή τη συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι σόφρον, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι δίκαιο. Συγγνώμη. Πρόεδρος. Συμφωνώ. Θα ήθελα να δώσω σε όλους χρόνο αγόρευσης. Δυστυχώ όμω υπάρχουν κάποιοι που θέλουν το λόγο και δεν είναι στον κατάλογο. Εσείς είστε στον κατάλογο και εγώ θα πρέπει να ιεραρχήσω και θα δώσω το λόγο και στου συναδέλφους στη διάρκεια της ε, διαδικασίας Catch the Eye. Δεν μπορώ όμως να δημιουργήσω πρόβλημα με τις υπηρεσίες. Δεν μπορώ να δώσω σε όλους το λόγο. Ελπίζω όταν σας δώσω το λόγο να μπορέσετε να πείτε αυτά που θέλετε. Σημειώνω όμως την παρατηρήσή σας. Ο κύριος Καβαντά για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί για πρώτη φορά σε μια Ήπειρο μια κοινοβουλευτική συνέλευση προσπαθεί να επανεξισορροπήσει τις σχέσεις μεταξύ γκάφα, αυτών των μεγάλων ε, ομίλων ε, και αυτών που τις τροφοδοτούν, δηλαδή δημιουργούσε και τύπο. Η δημιουργική κλάδη 130 δις ε, το χρόνο και 1.700.000 εργαζόμενοι στην Ευρώπη απειλείται από τις άδικους συσχετισμούς, τους οικονομικούς. Κάτι όμως ακόμα πιο επικίνδυνο, όχι τόσο άμεσα, είναι ότι καταραίει ο τύπος, ε, η σχετική βιομηχανία. Και κανένας δεν προσπάθησε να το σταματήσει αυτό. Ο τύπος, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι η βάση της δημοκρατίας. Όταν δεν θα έχουμε πλέον ελεύθερο τύπο, όταν δεν θα υπάρχει στο Google κανένας δημοσιογράφος, ούτε στο YouTube, ούτε στη Wikipedia, ούτε πουθενά άλλου, δεν θα έχουμε πλέον ενημέρωση, απλά μόνο φήμες σαν αυτές που ακούμε και κυκλοφορούν εδώ και ορισμένους μήνες. Αυτό το κείμενο είναι η μόνη ευκαιρία για τους δημιουργούς και για τις επιχειρήσεις του τύπου και τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους να πάνε επαναξισορροπήσουν προς όφελός τους και θα έλεγα να προστατεύσουν το μέλλον τους εξού και πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο και να το ψηφίσουμε συνολικά αρνούμενοι να δεχτούμε οποιαδήποτε τροπολογία. Το κείμενο αυτό πρέπει να το δούμε ως ένα πρώτο βήμα γιατί για να υπάρχει ξεσορρόπηση στην όλη κατάσταση χρειάζονται και άλλα βήματα. Γίνεται λόγος για λογοκρισία, για φιλτράρισμα, ε, για τη Wikipedia μας μιλάνε, η οποία προστατεύεται στο κείμενο. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν υπάρχει φιλτράρισμα. Γιατί όμως φτάσαν μέχρι εδώ στην Ολομέλεια αυτές οι ιδέες, γιατί για πρώτη φορά μέσα σε 15 χρόνια που είμαι ευρωβουλευτής μας βομβάρδισαν σαν να είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι, διανοούμενοι ε, τα ιερά τέρατα ε, της οικονομίας που θέλουν τις δραστηριότητές μας να τις φετεριστούν. Πρέπει να το ψηφίσουμε όλο αυτό το κείμενο συνολικά, γιατί αλλιώς ε, θα, αυτό θα έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις διακόπτη το μιλητής. Sorry, colleagues. Just to say... Πρόεδρος, 12 έχω ήδη στον κατάλογο και για το κατσιά και αυξάνει το αριθμό αυτό. Κύριε Ρέντε, τρεπτά κυρίε και κύριοι, Τρία πράγματα σε αυτή τη συζήτηση που άπτεται των πνευματικών διαματών είναι πρωτοφανή. Πρώτα απ' όλα, 200.000 άνθρωποι αυτό το Σαββατοκύριακο διαδήλωσαν κατά τη μεταρρύθμιση αυτή. 5 εκατομμύρια έχουν υπογράψει ένα petition κατά του upload filter, του φίλτρου αναφόρτωση. όμως ε, ε, δεν το έχει λάβει κανεί υπόψη, ε, υπόψη ότι Πρώτη φορά γίνεται τέτοια ε, αναστάτωση κατά μια οδηγίας της Ένωσης ε, και αγνοείται εντελώς αυτή η διαμαρτυρία. Ε, αντί όμως να υπάρχει κάποια κριτική, προσβάλλονται όσοι προσπαθούν να υψώσουν τη φωνή τους και έχουμε όπως ίσως και ο κύριος Καβαντά πιστεύει, πολλού να θεωρούν ότι τα email δεν τα στέλνουν οι εκλογείς στους βουλευτέ αλλά bots. Και η Κομισιόν λέει ότι είναι μία μάζα η, ε, αυτοί που ασκούν κριτική. Και το Τσέντε, ο υπεύθυνο θεωρεί ότι πληρώνονται αυτοί που ε, διαμαρτύρονται. Ε, όλα αυτά είναι δυσφήμιση που πολύ εύκολα μπορεί κανείς να την αντικρούσει και θεωρούν κάποιοι ε, ότι ε, τέλος πάντων αυτά τα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομάδες λόμπι και τα παρουσιάζουν ε, οι επιφυλίδες κάποιων εφημερίδων. Ε, θεωρούν ότι όλα αυτά κάποιοι προέρχονται από την Αμερική και έτσι δεν σκέφτονται επί της ουσίας ε, τι γίνεται. Δεν τους νοιάζει ε, που υπάρχουν προειδοποίησεις και από τον ίδιο τον Ομοσπονδιακό υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων σε ό,τι αφορά το upload filter και ο εκπρόσωπος για τα ελευθερία το γνώμης και πολύ σημαντικά ερευνητικά κέντρα για άλλα Όματα. Κανένας δεν θεωρεί ότι είναι σημαντική αυτή η μεταρρυθμίση τσέντε ούτε τεσπεντέ ούτε και αντιπολίτευση ε, και κανείς δεν θέλει να πάρει την πολιτική ευθύνη για το upload filter του άρθρου 13 όπου το θεωρούν όλοι κάτι ανόητο μέχρι και η κυρία Μέλκε παρακαλώ λοιπόν να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας παρακαλώ διακόπτω γιατί θέλω να ερεμήσουν κάποιοι συνάδελφοι που φωνασκούν Κύριε Μπροκ, Παρακαλώ. Έχει το λόγο η κυρία Ρέντα αυτή τη στιγμή. Να σεβόμαστε παρακαλώ τον ομιλητή που είναι στο μικρόφωνο. Κυρία Ρέντα, συνεχίστε. Κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη ε, στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ε, για το upload filter παρόλα αυτά ε, ψηφίζουν ε, στην ε, κυβέρνηση υπέρ και μάλιστα η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung έχει ανακαλύψει το ότι υπήρξε ένα παζάρ μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας δέχτηκαν οι Γάλλοι το upload filter για να ψηφίσει το Nord Stream η Γαλλία. Το πιο τραγικό, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, Χαίρομαι που έχετε ξυπνήσει όλοι έτσι πολύ καλά σήμερα. Το πρέπει παρακαλώ μην ακούτε από δεξιά από αριστερά φωνές. Το τραγικότερο είναι ότι η νέα γενιά που για πρώτη φορά θα ψηφίσει φέτος στις ευρωεκλογές ήδη μαθαίνει το μάθημά της. Δηλαδή τους λέμε δεν αξίζει τίποτα η διαμαρτυρία σας, οι πολιτικοί θα συνεχίσουν να ψεύδονται και δεν θα επηρεαστούν καθόλου ούτε από τα πραγματικά στοιχεία και τα επιχειρήματα αν ε, αυτά δεν προωθούν τα γεωπολιτικά του συμφέροντα. Αυτό, η αίσθηση αυτή της αδυναμίας θα τους στιγματίσει τους νέους μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να προχωράμε γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελευθερία του διαδικτύου αλλά και μια ολόκληρη γενιά θα τους ε, κλέψουμε αν θέλετε την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική και δεν είναι αυτό. Διακόπτεται η πρόεδρος. Πρέπει να καταψηφίσουμε το 13 λέει η κυρία. Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασπάρη έχει μια ερώτηση. Το δέχεστε? Το ερώτημα ναι το δέχομαι. Αξιότιμη συνάδελφε Ρέντα, ουσιαστικά ε, εμένα είπατε ότι είπα πως ε, είναι πληρωμένοι αυτοί που διαδηλώνουν. Να σας επαναλάβω ότι είπα ξεκάθαρα και σας παρακαλώ να ε, λαμβάνετε υπόψη αυτά που λέω εγώ και όχι αυτά τα οποία επίτηδες παρερμηνεύετε εσύ και η Είπα Εγώ ότι γίνεται δημοσία προσπάθεια ακόμη και με πληρωμένους διαλωτές να ε, μην προωθηθεί αυτή η οδηγία για την προστασία των Εγώ δεν μίλησα για τους νέους, για τις δισεκατομμύρια νέους και νέες οι οποίοι κατεβαίνουν. Διακόπτεται. Κύριε Κασπάρη, 30 δευτερόλεπτα είχατε για να κάνετε ε, μία ερώτηση. Αυτό που θέλετε να πείτε το είπατε. 30 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ο κανόνα. Και έτσι λειτουργούμε, με κανόνε εδώ. Κυρία Ρέντα θα απαντήσει τώρα. Κυρία Κασπάρη, μόνο σας ε, το είπατε ότι κάποιοι διαδηλωτές ήταν πληρωμένοι και μιλήσατε για 450 ευρώ. Σα ακούσαμε, σα ακούσαμε όλοι, είπατε για 350 ευρώ και ε, το έντρι για τα, ε, ο οργανισμός για τα δικαιώματα έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ ε, για να έχουν επαφές άσκησης πίεσης. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμως που πληρώνουν εδώ μόνοι τους τα τα οδηπορικά του. Θέλατε για διαδικαστικό κάποιο το λόγο. Λοιπόν, ένα λεπτό ε, έχετε χρόνο αγόρευση στη συνέχεια. Θέλετε τώρα μήπως να το χρησιμοποιήσετε το λεπτό σας. Εκτός μικροφώνου κάποιος φωνασκεί. Okay. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν με αφήνετε, φωνάζει κάποιος να υποβάλω ερώτηση. Ψεύδεται η συνάδελφος, ψεύδεται Ενώπιν της ολομελίας. Πρόεδρο, σα ακούω, αλλά δεν σα ακούν οι άλλοι, γιατί το μικρόφωνο σα δεν λειτουργεί. Κύριε Ρέντε, παρακαλώ, καθίστε. Εγώ ω πρόεδρο, θα φροντίσω όσοι προσήλθαν να έχουν χρόνο στο ΚΑΤΣΤΙΑΗ, Αλλά δεν μπορείτε να διακόπτετε την συνεδρίαση. Κύριε Ρέντα, θα δεχτείτε μία σύντομη ερώτηση του κύριου Ρέντε. Ωραία, 30 δευτερόλεπτα κύριε, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Σας ερωτώ λοιπόν, πού είναι το περίφημο φίλτρο αναφόρτωσης Πού είναι κυρία Ρέντα αυτό το upload filter συγκεκριμένα στο κείμενο πείτε μας πού είναι, πού το λέει. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. ότι με ρόντε, Λέει ότι οι πλατφόρμες ε, θα πρέπει να ε, μην επιτρέπουν ε, την αναφόρτωση κατοχυρωμένων πραγματικά δικαιώματα και δεν χρειάζεται να έχουν κάποια άδεια. Και λέει εκεί ότι μπορούν να έχουν αυτό το upload filter, αυτό το φίλτρο, να γίνει αυτό το φιλτράρισμα αναφόρτωσης. Please, colleagues. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Σμαστάλκα. 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συνεδρίαση μοιάζει μάλλον με τελικό παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Δεν μοιάζει με κοινοβουλευτική συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μιλώ εξ όλων. Αν ε, λέω ότι θα είμαστε όλοι ανακουφισμένοι όταν υπερψηφιστεί το κείμενο. Αλλά και αν δεν ψηφιστεί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έχουμε τα άρθρα 11 και 13, τα πιο επίμαχα, τα πιο αμφιλεγόμενα. Κοιτάξτε, μετά από ένα μισό χρόνο δεν είμαι ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα. Εγώ θα είμαι κατά τη πρόταση. Πάντω, σπαταλήσαμε μια εξαιρετική ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε τον χώρο της πνευματική ιδιοκτησίας και να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανταυτού, έχουμε μια πρόταση η οποία εξαπαρά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εισάγει λογοκρισία, ευνοεί τα chat και εν τέλει ευνοεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα είναι το τέλος του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Επιπλέον πιστεύω ότι εάν υπερψηφίσουμε τη σημερινή έκθεση, αυτό θα είναι χαστούκι στο πρόσωπο εκατομμύριων ανθρώπων που μας στέλνουν ε, email ε, και διαμαρτύρονται στους δρόμους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, πρέπει να κάνει κάτι για να μην χάσει την αξιοπιστία του. Τέλος πια στην υπεροψία. Να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά, Μας πιέζουν και δύο πλευρέ. Από τη μια πλευρά ακούμε για χιλιάδε ανθρώπων που ανησυχούν για το μέλλον του ίντερνετ και από την άλλη έχουμε ακριβέ δεξιώσει ε, υπέρ του κειμένου. Μην νομίζετε πάντως ότι οι δημιουργοί στηρίζουν την πρόταση. Οι μεγάλοι παίκτες την υποστηρίζουν. Εμένα όμως με ενδιαφέρουν οι ψηφοφόροι μου, οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια να χρησιμοποιούν λόμπιστ. Ε, Τι χρειαζόμαστε, μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δημιουργών και από την άλλη μεριά ε, της προστασίας των καθημερινών απλών ανθρώπων. Η προτινόμενη νομοθεσία, ειδικά με τα άρθρα 11 και 13, δεν πετυχαίνει αυτήν την ισορροπία. Πρόκειται για ανελεύθερο μέτρο, διότι στην πράξη οι μεγάλες εταιρείε θα χρησιμοποιούν τους πολίτες ως ε, αυτομάτως ενόχους. Θα σταματήσει το περιεχόμενο να αφαιρείται αυτομάτως. Έτσι, ισοπεδώνοντας τα πάντα, γνώμη τους εθνικούς κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Πρόκειται για ναρκοπαίδιο. Εν τέλει, το νόμιμο περιεχόμενο θα αντιμετωπίζεται ως παράνομο. Τι βλέπω λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον, η γνώμη των ε, Βρετανών που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αλλάξει. όσο και το αντίθετο. Πού πηγαίνουμε. Φοβούμαι ότι κάποιοι που ήταν υπέρ τη παραμονή τώρα θα ψηφίσουν Brexit λόγω αυτής της νομοθεσίας. Λοιπόν, με την πρόταση αυτή απομακρύνουμε τους νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κακή νομοθεσία. Είναι δυστυχώς νομοθεσία της τελευταίας στιγμής. Μετά από μισή εβδομάδε εμεί θα έχουμε κλείσει την ε, θητεία μα. Λοιπόν, α μην βιαστούμε για άλλη μια φορά. Δυστυχώ δεν λάβαμε υπόψη μα αυτά που έπρεπε να λάβουμε υπόψη μα. Ακούστε, αφουγκραστείτε του ψηφοφόρου σα. Α έρθουμε πιο κοντά στον Βρετανικό λαό, στο λαό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπλε κάρτα. Το κύριο Στρογεύσκη, την δέχεστε. Κύριε Στρογεύσκη, 30 δευτερόλεπτα. Είμαι ένας από τους τελευταίους ε, που στέσονται με τα λόμπι, όμως θα ήθελα να ξεχωρίσουμε τα διαφορετικά λόμπι. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα για το δικαίωμά τους στην αμοιβή. Η ερώτησή μου προς σας, κυρία, είναι δεν βλέπετε ότι υπάρχουν τα μεγάλα εμπορικά λόμπι οι γίγαντες της αγοράς και οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι απλώς διεκδικούν την αμοιβή τους. Ευχαριστώ. Καμία αντίρρηση να αμείβονται αυτοί που πρέπει να αμείβονται. Και καλώς υπεραμείνονται του δικαιώματός τους. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, επαναλαμβάνω. Καμία αντίρρηση. Όμως, ξανά και ξανά τη βλέπουμε τα μεγάλα συμφέροντα, αυτά που μας πιέζουν, παρά οι δημιουργοί. Οι δημιουργοί στη δική μου εκλογική περιφέρεια λένε ότι δεν του ακούμε. Αν και εν τέλει κανείς δεν θέλει αυτή την νομοθεσία. Οι απλοί πολίτες ανησυχούν με το άρθρο 11 και 13. Πρόεδρο, και από τον λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σήμερα ε, ασχολούμαστε με την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι μία ιστορική ημέρα ή μία μαύρη ημέρα αντίθετα. Είναι απότοκη ε, τριετούς εργασίας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση ίσα ίσα ε, σφετερίστηκε το όλο ζήτημα η Silicon Valley. Δεν υπερασπιζόμαστε τους δημιουργούς και χρήστες. Οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιγραμμικές ε, πλατφόρμες που πολλές φορές αποσύρουν τα, το περιεχόμενο. Οι δημιουργοί έχουν δικαίωμα ίσης και δίκαιης αμοιβή. Ο Μαλρό έλεγε ότι ότι ο πολιτισμός δεν κληρονομείται, κατακτάται. Ο Σκιώδης λοιπόν λέω ναι στον πολιτισμό, ναι στα δικαιώματα των ε, δημιουργών, των εκδοτών και των καλλιτεχνών. Ο κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και ειδικά στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζουν λογοκρισία βασισμένη αποκλειστικά στι επιθυμίε και τα συμφέροντα των ιδιοκτητών του. πώ άραγε νομιμοποιούνται οι ιδιωτικοί φορεί να περιορίζουν θεμελιώδει ελευθερίε; οι σημάνσει και η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιούνται ω εργαλείο στιγματισμού ή εξοβελισμού ανεπιθύμητων ή ανταγωνιστικών ιδεών και προσώπων. για παράδειγμα μόνο η απλή αναφορά του ονόματό μου ή κοινοποίηση ομιλία μου στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σε συγκεκριμένο μέσο κοινωνική δικτύωση, αρκεί ώστε να τιμωρηθεί ο κάτοχος του λογαριασμού με ποινή αποκλεισμού για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ή να του κλείσουν το προφίλ. εάν λοιπόν σε αυτό το ήδη ζωφερό για την ελευθερία του λόγου περιβάλλον προσθέσουμε και ορουελικής εμπνεύσεω λογισμικά που θα ανοιχνεύουν τι απαγορευμένε λέξει. καταλαβαίνουμε πω θέτουμε τι βάσει για μια καταπίεση των ελευθεριών βγαλμένη από τι πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας που αρμόζουν μόνο σε σοβιετικά καθεστώτα. σας ερωτώ λοιπόν αυτό είναι το μέλλον που επιθυμείτε για την ένωση; εμείς σίγουρα όχι και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση και κυρίως τη συγκεκριμένη διάταξη. ευχαριστώ. Η κυρία Φερχάιν για 1,5 λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, εδώ και πάνω από δυόμιση χρόνια στο Κοινοβούλιο τσακωνόμαστε με τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμβιβαστική πρόταση. Και έχουμε ένα κείμενο επιτέλου ε, που θα οδηγήσει σε περισσότερη δικαιοσύνη στο διαδίκτυο και θα αναλάβουν τι ευθύνε του και οι μεγάλοι όμιλοι. Σίγουρα είναι δικαίωμα βασικό η προστασία των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, να προστατευτούν τα έργα των δημιουργών κοινωνία μας ε, δεν έχει στόχο ε, να μην προστατεύουμε. Θέλουμε κατά ε, ελάχιστα εισοδήματα και άλλα βασικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να βάζουμε, να μην βάλουμε εμπόδια στους μεγάλους ομίλους για να ζητάνε αστρονομικά ποσά και να κερδοσκοπούν σε βάρος των δημιουργών. Έχουμε λοιπόν πιο απλές διαδικασίες αδειοδότησης ε, ε, στο 70, στο 17, στο 7, στο 9. Ε, θέλουμε την κατοχήρωση της ελευθερίας έκφρασης. Υπήρχαν κάποιες δυσανάλογες διατάξεις, ε, τις οποίες ε, τις έχουμε απαλείψει. Dropbox, eBay, ε, Wikipedia δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία και επίσης ρυθμίζουμε τα όσα ισχύουν για τους μικρούς εκδότες και για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι αναλογικά λοιπόν τα μέτρα και θέλουμε δικαιοσύνη στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες είναι αυτές οι οποίες ε, ε, έχουν το περισσότερο κέρδος. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη, δεν θέλουμε άναρχο καπιταλισμό όπως αυτός που βιώνουμε εδώ. Θέλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον άναρχο καπιταλισμό. For one minute, Madam Η κυρία Ροζιέρ για ένα λεπτά. Ευχαριστώ. Η οδηγία είναι απότοκη μια εργασίας δυόμιση ετών δημιουργεί εκδότες, δημοσιογράφοι, ερευνητές ε, έχουν συμμετάσχει, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι ίδιοι οι χρήστες γιατί θα μας δώσει την ασφάλεια δικαίου που θέλουμε και δεν θα είναι αυθαίρετες πια οι πλατφόρμες. Έτσι η Ευρώπη ε, θα μπορέσει να είναι κυρίαρχη σε σχέση με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις που λαιλατούν τα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτική μας ζωή και καταπατούν τα δικαιώματα των δημιουργών. Πώς ε, είναι δυνατόν να μην αμείβεται η εργασία γιατί είναι σε ψηφιακό πλαίσιο. Όλοι πρέπει να αμείβονται. Τα μεγάλα ε, λόμπι ψεύδονται. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις παραβιάσεις διαφάνειας και πολλές φορές υπάρχει σκιώδης χρηματοδότηση πλατφόρμων. Ελπίζω λοιπόν να σταθούμε κατά του άκρα του νεοφιλελευθερισμού και υπέρ των Ευρωπαίων Χριστών. Ο κύριος Λοσλοτόφσκι για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικά χρόνια πριν ε, έγινε ε, μία, υπήρξε μία διχογνωμία για το τι μας απασχολεί εδώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της οδηγίας είναι το γεγονός ότι η ερμηνεία θα είναι πιο σοβαρό ζήτημα από το ίδιο το κείμενο. Ο κύριος Βος δεν μας έπεισε με την ε, παρουσίασή του. Δυστυχώς οι ορισμοί δεν είναι συγκεκριμένοι ε, και γι' αυτό ακριβώς θα υπάρξουν πολλά κενά και στη δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς ε, οι κολοσσοί ορίζουν τη δημόσια συζήτηση και τη μονοπολούν. Και γι' αυτό θα ήθελα να καταψηφίσετε αυτή την οδηγία. Ρόντε για ένα λεπτό. Κύριε, κύριε Ρόντε. Πραγματικά είναι απίστευτο το ότι εδώ σήμερα ακούμε ε, την αριστερά να λέει πράγματα που κανονικά δεν λέει ε, η αριστερά. Ε, δεν υπάρχει για να καταρρύψω, καταρρύψω κάποιους μύθους ε, δεν υπάρχει αναφορά στο upload filter δεν υπάρχουν φίλτρα ε, ε ούτε περιορίζονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών αντιθέτως ελέγχεται κάπως η κατάσταση με τις πλατφόρμες το facebook και άλλοι γιγαντές δεχόμαστε σήμερα πολύ ε, ελαφρά την καρδία ε, να επηρεάζουν το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί ε, να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ενώ οι δημιουργοί δεν έχουν ούτε δικαιώματα, ούτε ελέγχουν τα δικά τους ουσιαστικά δημιουργήματα. Και Πραγματικά αυτή η κολοσσοί της τεχνολογίας που δεν πληρώνουν μισθούς, που δεν πληρώνουν φόρους, είναι ανεξέλεγκτη. Και έτσι φτωχαίνουμε και οικονομικά και πολιτισμικά. Ελπίζω να στηρίξετε σήμερα το... Κυρία Τρούπελ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλουμε ελεύθερο αλλά και επιτέλους δίκαιο ίντερνετ. Δεν θέλουμε ανευθυνότητα. Δεν θέλουμε όμως ούτε και λογοκρισία. Ε, στην Κίνα υπάρξει, υπάρχει λοκρισία, δεν υπάρχει προστασία πνευματική συντοξία. Αυτό που θέλουμε είναι οι ενεργέ ε, πλατφόρμε περιεχομένου να έχουν άδεια. Ε, και έτσι θα είναι όλοι κερδισμένοι. Αυτό που θα αναφορτώνει θα έχει κάποια δικαιώματα και οι πλατφόρμε θα παίρνουν την ευθύνη επιτέλου και θα υπάρχει και μια αναλογική αμοιβή για το δημιουργό. Αυτό θα φέρει δικαιοσύνη στο ελεύθερο διαδίκτυο, κάτι που όλοι επιθυμούμε. Χρειάζονται γενικοί κανόνε ε, για τον καπιταλισμό των πλατφορμών. Πρέπει να πληρώνουν φόρου και να λαμβάνουν ευθύνε ε, όταν κάνουν εκστρατεία πληροφόρηση. Θέλουμε την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και δεν μιλάμε για υπερρύθμιση εδώ, αλλά για δίκαιους κανόνες, γιατί ε, είναι οι ε, κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων η μειοψηφία στην κοινωνία μας και χρειάζονται την προστασία μας. Ψηφίστε παρακαλώ το κείμενο αυτό, γιατί θα φέρει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Μίχελς. Βλέπω να χαιρετίζεται ορισμένη την εναρμόνιση ε, στα πνευματικά δικαιώματα. Όμως αυτοί που είναι υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης ε, ε, λένε ότι ενισχύεται ο δημιουργικός κλάδος. 5 εκατομμύρια άνθρωποι όμως και σας παρακαλώ και αυτοί είναι δημιουργοί, έχουν υπογράψει αυτή την αναφορά. Δεν θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα οι μηχανές. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος δικαίου και αυτό το ε, άρθρο 13 ή 17 ε, γίνεται λόγος για αυτό το upload filter. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η διάταξη για τις αδειοδοτήσεις. Η ρύθμιση των πλατφορμών πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Ψηφιακό φόρο, ηθική αλγόριθμη, έλεγχος των καρτέλ ε, και καταπολέμηση των μονοπωλίων. Ας βρούμε λοιπόν καλύτερες λύσεις ε, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε ελεύθερη επικοινωνία τον 21ο αιώνα και όχι εκαθάριση στο διαδίκτυο ότι δεν μας αρέσει. Mr. one Είμαστε υπέρ της προστασίας των δημιουργών. Η οδηγία δυστυχώς προάγει τα συμφέροντα των πολυεθνικών, αυξάνει τα κέρδη τους. Έχει σκοπό να καταπνίξει τον ελεύθερο λόγο, τη διαφορετική άποψη. Αυτό θέλουν τα καθεστώτα. Οι διαφορετικές φωνές ήδη αποκλείονται από τις πλατφόρμες. Αυτό κάνουμε ακριβώς με την οδηγία. Θεσμοθετούμε την λογοκρισία. Επ' αυτού ψηφίζουμε. Οι βουλευτές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε σύντομα εκλογές. Οι ψηφοφόροι να σημειώσουν ποιοι υπερψήφισαν και ποιοι καταψήφισαν αυτήν την οδηγία και να καταψηφίσουν αντιστοίχως τον Μάιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μαζί με τους μεγάλους παίκτες να καταπνίξουν τις ελεύθερες φωνές. Ε, αυτοί οι βουλευτές που θα υπερψηφίσουν αξίζει να χάσουν τη θέση τους στο Κοινοβούλιο. είναι ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, χάρη στη συνεισφορά όλων, το διαδίκτυο είναι μια μικρογραφία του κόσμου μας. Σα συνοχλεί. Δεν θέλουμε υπερβολική νομοθέτηση. Το διαδίκτυο είναι το τελευταίο προπύργιο ελευθερίας και γι' αυτό κάποιοι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό δείχνει ότι οι κανόνες σας είναι βλαβεροί θα ήμασταν καλύτεροι χωρί αυτού του κανόνε. Αυτό είναι το διαδίκτυο, η ελευθερία. Χωρί του κανόνε αυτού θα είχαμε μια καλύτερη ζωή. Αυτήν προσπαθείτε να καταστρέψετε. Όποτε και όπω μπορείτε. Λοιπόν, όχι, δεν θα σα αφήσουμε να θέσετε τροχοπέδι στη ζωή, την ελεύθερη ζωή των ανθρώπων. Δεν θέλουμε τις παγίδες που προσπαθείτε να δημιουργήσετε στο διαδίκτυο. Δεν Grandes Πασκουάλ για ένα λεπτό. Το περίφημο άρθρο 13 προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για το τι θα κάνουν οι πλατφόρμες τη στιγμή που δεν προασπίζονται τα δικαιώματα των ε, δημιουργών. Και αυτό αφορά και τον τελικό χρήστη. Δηλαδή, ε, το περιεχόμενο θα πρέπει να την χάνει προστασίες γιατί την πνευματική ιδιοκτησία την κατέχουν οι δημιουργοί, είτε είναι υλικό είτε άϊλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπερασπιζόμαστε το περιεχόμενο των δημιουργών. Υπάρχει πνευματικό, πνευματική δημιουργία, γιατί η πλατφόρμα είναι αυτή που ευεργετείται από το περιεχόμενο μέσω διαφημίσεων η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την αδειοδότηση έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να καταλυστεύει το περιεχόμενο χωρίς τη θετική γνώμη των δημιουργών. Αυτό ακριβώς είπαμε και στους τριμερείς διαλόγους. Νομίζω ότι θα πρέπει να τύχει της υποστήριξής μας αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέλκιν για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μόνο η Google είναι κατά της μεταρρύθμισης, λένε αυτοί που είναι υπέρ της οδηγίας. Δεν ισχύει όμως αυτό. Ε, και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μάλλον για τα προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και πολλοί άλλοι θεωρούν ότι τελικά ε, οι ε, φορείς διαχείρισης θα ισχυροποιηθούν. Όχι όμως οι δημιουργοί, γιατί τελικά πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από την πνευματική δοξία, αλλά με τη δημοκρατία μας έχει να κάνει. 5 εκατομμύρια υπογράφουν αυτή την petition και τους λένε ότι είναι ένα, μια μία μάζα ε, από την Κομισιόνα ε, και πολλοί ε, θεωρούν ότι αυτοί οι οποίοι είναι κατά δεν εκφράζουν τις γνώμες τους αλλά το έκαναν κάποια bot, κάποιες μηχανές το διαδίκτυο ή ότι κάποιοι για να κατέβουν ε, στο δρόμο να διαδηλώσουν έχουν πάρει 450 ευρώ. Επομένω, πλήττεται τη δημοκρατία μα. Πρέπει ιδίω του νέου Ευρωπαίου να του λάβουμε σοβαρά υπόψη, οι οποίοι θέλουν ε, να παραμείνει το ίντερνετ όπω το θέλουν, γιατί με το άρθρο το 13 και με το κείμενο αυτό καταστρέφεται το διαδίκτυο όπω το θέλουν. Πρέπει λοιπόν να διαγράψουμε το άρθρο 13. Ευχαριστώ. Κύριε Βέλκεν, έχετε από τον κύριο Ράτκερ μία μπλε κάρτα. Ναι, αγαπητέ ε, συνάδελφοι, ε, μας είπες ε, πόσοι άλλοι εκτό του Google είναι κατά η υπουργό δικαιοσύνη, η κυρία Μπάλα από το S5 δεν ήταν μεταξύ αυτών που αναφέρατε, την ξεχάσατε. Ψήφισε στο Συμβούλιο υπέρα, αλλά τώρα λέει όχι πρέπει να ψηφίσουμε κατά. Άρα δεν τα έχουμε πολύ καταλάβει. Μήπω πρέπει να μα εξηγήσετε τι συμβαίνει. Αγαπητέ Ντένι, ε, τιμή μου να σε βοηθήσω να καταλάβεις. Ε, η ε, υπουργό δικαιοσύνη ε, ήταν κατά και ουσιαστικά έπρεπε να τηρήσει τη συμφωνία μεταξύ Μέρκελ και Γαλλίας που κατήγγειλε χθε η ΕΦΑΤΣΕΤ. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν. Ο κύριος Λούκε για ένα λεπτό έχει το λόγο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 Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ε, είναι απίστευτο αυτό το οποίο αποκάλυψε η ΦΑΤΣ, ε, η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Γίνονται παζαρέματα από τη μία το upload filter και από την άλλη ο Nord Stream. Ε, δεν είναι έτσι η πολιτική όμως. Κανονικά θέλουμε αντικειμενικότητα. Πρέπει να δούμε αν χρειάζεται τελικά αυτό το φιλτράρισμα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής θυξίας. Κανείς δεν θέλει να στερεί το εισόδημά τους από τους δημιουργού. Τι κάνουμε κάνουμε όμως με αυτά τα φίλτρα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και αν θεωρούμε ε, και λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχει αναφορά σε αυτά τα φίλτρα, σε αυτό το κείμενο, αυτό είναι αναλυθές. Πριν ε, δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο, οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν ε, πρώτα επαληθεύσει κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι φίλτερο. Είναι δηλαδή απλό φίλτερ μέσα στην ε, οδηγία. Ε, και υπάρχουν κάποιοι μικροί ε, ε, Φορεί εδώ, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Το άρθρο 13 πρέπει να διαγραφεί από την οδηγία ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ψηφίσουμε για την προστασία των δικαιωμάτων τη Ευχαριστώ για να την κυρία Τούμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συναδελφοί. Το ότι χρειάστηκαν δυόμιση χρόνια για αυτήν την οδηγία δεν την κάνει δυστυχώς καλύτερη οι επιπτώσει στα δικαιώματα του ανθρώπου είναι πολύ σοβαρέ και το λένε πανεπιστημιακοί, ΜΚΟ, καθώ και ο ειδικό ε, για τα δικαιώματα του ανθρώπου από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αν διαβάσουμε την ε, Οικουμενική Διακήρυξη, όλοι έχουν δικαίωμα στην πληροφορία μέσω οποιοδήποτε καναλιού, φορέα κλπ. Και αυτό ακριβώς καταργούν τα άρθρα 11 και 13. Δημιουργούν εμπόδια στην κυκλοφορία τη πληροφορία. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημιουργών. Ναι, όμως ε, εκεί έχουμε πολύ διαφορετικούς παίκτε. Δεν είναι ισόρροπη η πρόταση. Δυστυχώ, εδώ βάζουμε μπροστά τα συμφέροντα των λίγων. Τον Σεπτέμβριο είχαμε πολλέ εναλλακτικέ μπροστά μα στο τραπέζι και σήμερα όχι πια δυστυχώς. Οπότε θα καταργήσουμε τα 11 και 13 ή θα καταψηφίσουμε. Γιατί αλλιώ το πλήγμα κατά τον δικαιωμάτων του ανθρώπου θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άντερσον, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο λόγια για την γελία θεωρία συνωμοσία του λόμπι του copyright. Εμείς θέλουμε ένα ελεύθερο διαδίκτυο. Δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα του Google και του Facebook. Συγγνώμη, η θεωρία συνωμοσία είναι για τα σκουπίδια. Δίνουμε μάχη κατά αυτών των γιγάντων εδώ και χρόνια. Δίνουμε μάχη για την ιδιωτικότητα, δίνουμε μάχη κατά των μονοπωλίων. Εγώ θα ήθελα να χτυπήσουμε την Google και το Facebook εκεί που τους πονάει να, ψηφίσουν, να πληρώσουν φόρους Γι' αυτό να δώσουμε αγώνα. Να δώσουμε αγώνα για την ιδιωτικότητα, να δώσουμε μάχη για την ανέλεψη ευθύνη. Όμω, εδώ πρόκειται για τη λάθο μάχη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι το Google και το Facebook, αλλά εμπιστεύομαι του ειδικού που λένε ότι τα άρθρα 11 και 13 είναι κάκα για το διαδίκτυο και ότι δεν πρέπει να πέσουν θύματα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι καιρός να νομοθετήσουμε για να περιορίσουμε τους γίγαντες της Βορειοαμερικής, να βάλουμε ένα φρένο, να πληρώσουν αυτοί οι μεγάλοι τους δημιουργούς. Κατανοώ τις πιέσεις των γιγάντων του κλάδου, όπως το υπενθύμισε ο κύριος Καβαντά. Μιλάμε για 536 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πιο πολλοί δουλεύουν στις μέρες μας ε, στη δημιουργία δημιουργικού παρά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την πολιτισμική πολυμορφία, για τον πλουραλισμό. Η οδηγία υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να δείξουν σεβασμό προς τους δημοσιογράφους, προς τους δημιουργούς παρέχοντας και νομική ασφάλεια η οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Εγγυάται δικαιώματα και ευνοεί την πρόσβαση στη γνώση προάγει τα δικαιώματα των δημιουργών. Προστατεύει τους δημιουργούς. Αυτό ακριβώς προστατεύουμε και εμείς τη δημιουργία ε, εκ μέρους των δημιουργών. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σόλτεκ για ένα λεπτό. Αυτή η εκδοχή της οδηγίας εισαγάγει λογοκρισία, ένα επίπεδο λογοκρισίας που δεν είχαμε στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Δείτε τι λέει το κείμενο το ίδιο. Δεν μπορείτε να πείσετε τα μέλη εδώ όλοι έχουν οχυρωθεί πίσω από τις θέσεις τους ε, πολίτες της Ευρώπης. Εάν δεν θέλετε να χάσετε τις ελευθερίες σας, τότε θα πρέπει να πείσετε τις κυβερνήσεις σας ίσως να ε, αποχωρήσουν. Θα έπρεπε να πείσετε τις κυβερνήσεις σας να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε, ας εγκαταλείψουμε αυτό το γραφειοκρατικό τέρας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δημιουργήσουμε μία πραγματική ένωση των εθνών. Μία καινοτόμα ένωση των εθνών. Τι σας σταματάει από την καταψήφιση αυτού του κειμένου. Υπάρχει μία μπλε κάρτα. Θα δεχτείτε την μπλε κάρτα του κυρίου Στρογεύσκη. Δέχεστε την ερώτηση του κυρίου Στρογεύσκη. Τη δέχεστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε κύριε ότι ε, αντιτίθεστε σε αυτή την οδηγία, άρα να μην αμείβονται οι ε, δημιουργεί. Εσείς ε, είσαστε υπέρ ενός κόμματος που στοχεύει στην αποχώρηση έτσι ώστε η χώρα μας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και άλλη ε, μπλε κάρτα. Ο κύριος Καβαντά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα ο συνάδελφος ο οποίος ε, μας πείθει, θέλει να μας πείσει να αποχωρήσει από την να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε γιατί αυτός παρίσταται εδώ όταν του δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μικρόφωνο. Απάντηση με μικρόφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ναι, βεβαίως έρχομαι εδώ και ε, ε, δημοσία τάσομαι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θεωρώ ότι και άλλες χώρες θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σχηματίσουν μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση όχι ε, αυτό το γραφειοκρατικό τέρας, να δημιουργηθεί μία νέα Ευρωπαϊκή Ένωση καινοτόμα. Αυτό θα ήθελα να επισυμβεί για την Πολωνία ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θεωρώ ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάξει στάση, τότε θα πρέπει να αποχωρήσουμε και αυτό αφορά και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν περάσει πολλοί νόμοι και νομοθεσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η θέση μου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, απαντήσατε σε μία ερώτηση από τις δύο, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Άξελ Βός για την εξαιρετική του εργασία μέχρι τούδε. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες μάχες της τρέχουσας θητείας, γιατί Ευρώπη σημαίνει δημιουργία, εργασία και τέχνη. Πρόκειται για μία μάχη υπέρ της Ευρώπης. Ακριβώς για τι προασπίζομαστε αυτές τις αξίες. Αυτοί που καταφέρονται κατά τις οδηγίες θα πρέπει να δουν τι κάνουν οι πλατφόρμες. Εάν θέλουν να εισπράξουν δις δολάρια, θα πρέπει τότε να αναγνωρίσουν την εργασία του δημιουργού που τους επιτρέπει αυτά τα έσοδα. Δηλαδή στο Google να υπάρχει Φυσικά να υπάρχουν διαφημίσεις, αλλά να αμείβονται οι δημιουργοί. Ε, κύριε Ρέντα, μιλήσατε για νέους. Υπάρχουν νέοι που πληρώνονται 3 ευρώ το κομμάτι για την εξαιρετική τους δημοσιογραφία. Εάν θέλετε να τους υπερασπιστείτε, να υπερασπιστείτε το copyright. Για ένα λεπτό ο κύριος Γραμματικάκης έχει το λόγο η μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα ξεκίνησε ως μια τεχνική συζήτηση στην πορεία όμως εξελίχθηκε σε μάχη για την ψυχή της ευρώπης δηλαδή τον πολιτισμό και τις αξίες της. η συμφωνία δεν εξασφαλίζει μόνο ότι οι καλλιτέχνε και οι δημιουργοί θα επιβιώσουν στην ψηφιακή εποχή αποδεικνύει επίσης κάτι σοβαρότερο ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις δυνατότητές τους να παραπλανούν πολίτες και πολιτικούς και εντυπωσιάζομαι από το ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό. μετά από δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων λοιπόν και τρεις διαφορετικές επιτροπές πέντε και τρεις ψηφοφορίες στην ολομέλεια έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η οδηγία υποστηρίζεται από όλους τους επίσημους φορείς που πολύ την έχουν συζητήσει δημιουργών και καλλιτεχνών. Ως συζητής του Σοσιαλιστών στην Επιτροπή Πολιτισμού θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω όλους τους συναδέλφους που τάσσονται υπέρ του ανοιχτού και ελεύθερου διαδικτύου και δίκαιου όμως διαδικτύου να στηρίξουν το αποτέλεσμα του τριλόγου δεν θα είναι μια μάχη μόνο για το παρόν της ευρώπης αλλά επίσης αγαπητοί συνάδελφοι και για το μέλλον της. Ένα λεπτό κύριο Σούλικ. Ευχαριστώ πολύ. Η οδηγία, η τρέχουσα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα θα ε, αλλάξει επιταχύρω, ε, ιδίως ό,τι αφορά το άρθρο 13 με τη νέα αυτή πρόταση και το ίδιο θα γίνει και με το άρθρο 11. Ουσιαστικά θα περιλαμβάνονται και τα πολύ μικρά αυτά αποσπάσματα, παραθέματα που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο τι σημαίνει αυτό. Κοινωνικέ πλατφόρμες είναι αυτές που θα εξασφαλίζουν ε, την αποτροπή κλοπής περιεχομένου Δηλαδή αυτός που έχει ένα χώρο στάθμευσης, πάρκινγκ, θα είναι υπεύθυνο για το ενδεχόμενο κλοπής ε, κάποιου αυτοκινήτου ή απώλειας αντικειμένου μέσα από το αυτοκίνητο. Εκπλήσωμε επίσης ε, που δεν λαμβάνει υπόψη τη την κοινή γνώμη κομισιών. Για τα 11 και 13 έχω υποβάλει ε, τροπολογίες διαγραφής. Ευχαριστώ. Μπόγκοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όλοι έχουμε το δικαίωμα ε, της ελευθερίας έκφρασης. Μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στο διαδίκτυο, αλλά έχουμε και το δικαίωμα ε, της προστασίας. Θέλουμε ψηφιακό περιεχόμενο, ε, θέλουμε πνευματικά δικαιώματα, θέλουμε ελευθεροτυπία. Αλλά Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των δύο κατηγοριών δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει. Ο Άξελ Φως έκανε πολύ καλή δουλειά. Εστιάζουμε ουσιαστικά στους ε, μεγαλύτερους κολοσσούς ε, του διαδικτύου, πλατφόρμες που αποκομίζουν ε, τεράστιο κέρδος, αλλά δεν μοιράζονται το κέρδος αυτό με τους δημιουργούς. Αν θέλουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, και ανεξάρτητους ε, δημιουργούς γενικώ και καλλιτέχνες θα πρέπει να την εγκρίνουμε την πρόταση αυτή. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους μεγάλους αυτούς ε, ομίλους, ε, αλλά θα προστατεύσουμε τη δημιουργία. Θα στηρίξω λοιπόν την έκθεση αυτή, γιατί θα προωθεί στην ισότητα. Ευχαριστώ κύριο Μπλάνκο Λόπεθ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κανένας δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ανελευθερία στο διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς νόμους, αλλά δημιουργία υπάρχει μόνο αν υπάρχει δίκαιη αμοιβή. Αυτή η οδηγία προσπαθεί να διορθώσει αυτές τις ανισορροπίες για να ενισχύσει τους δημιουργούς, να δώσει χώρο στη αλυσίδα αξιών. Δεν καταλαβαίνω πώς ε, πολλοί εκπρόσωποι της αριστεράς δεν δέχονται τον πλούτο των πλατφορμών λέγοντας ότι υπερασπίζονται τους δημιουργούς. Δεν υπάρχουν ούτε μέμ ούτε hyperlinks. Αυτό αυτό είναι το διαδίκτυο του 21ου αιώνα. Είναι η ελευθερία του εκφράζεστε, η ελευθερία δημιουργίας και η σωστή αμοιβή των δημιουργών. Κύριε Μπλάνκο Λόπεθ, έχετε δύο μπλε κάρτες. Τις δέχεστε? Ο κύριος Ρούμπιχ και η κυρία Ματίας θα υποβάλουν την ερώτησή τους σε 32. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπλάνκο Λόπεθ κατά πόσον ισχύει ότι στο μέλλον ε, όταν κάποιοι αναφορτώνουν δεν θα έχουν ευθύνη όλοι ουσιαστικά όσοι δεν είναι επιχειρηματικοί. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο που είπε ότι δεν υπάρχει δημιουργία, αν δεν υπάρχει σωστή αμοιβή, θα ήθελα να διαβάσει την οδηγία εκεί που λέγεται ότι θα υπάρχει δίκαιη αμοιβή για τους ε, δημιουργούς. Εγώ δεν το βλέπω πουθενά αυτού. Πείτε μου πού αναφέρεται η δίκαιη αμοιβή για τους δημιουργούς. Βρείτε μου το παράθεμα. Μη λέτε λόγια θα πρέπει να επανισορροπήσουμε την αλυσίδα αξιών. Οι πλατφόρμες συνεισφέρουν για την δίκαιη αμοιβή, δηλαδή ανταμείβεται η εργασία, η δημιουργία δεν την χάνει εκμετάλλευση. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αριστερά θέλει να ευεργετούνται μόνο λίγοι ε, σε σχέση με τους δημιουργούς της Ευρώπης μας, των χωρών μας. Δεν είμαι σίγουρη ότι απαντήσατε στον κύριο Ρούμπιχ. Κύριε Μπλάνκο Λόπεθ, σας ε, υπέβαλε ερώτηση και ο κύριος Ρούμπιχ. Δεν απαντήσατε. Υπέβαλε την ερώτηση. Θυμόσαστε τι σας ρώτησε ο κύριος Ρούμπιχ. Κύριε Ρούμπιχ, μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπλάνκο Λόπεθ κατά πόσον ισχύει ότι οι χρήστε μα επαγγελματικοί δεν έχουν πλέον ε, κάποια ευθύνη ε, και ε, επομένω δεν μπορούν να, να, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια προσβολή για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία για το περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται σε κάποια πλατφόρμα από απλού χρήστε. Δεν είναι επαγγελματικοί. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων των μερών. Για τον αθλητισμό όμω, το ότι δεν συμπεριελήφθη δική μνήμα στα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών διοργανώσεων είναι κακό. Είχαμε το τροπολογία στο αρχικό άρθρο 12. 400 ψήφισαν υπέρ την προηγούμενη ε, Ολομέλη του Σεπτεμβρίου για αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να είχε υπάρξει μια τολική σκέψη ε, για την απόφαση Premier League Marfin ε, που σημαίνει θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η προστασία των αθλητικών διοργανώσεων από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα ανέλυε τα σχετικά συστήματα προστασία. Τελικά η επιλογή είναι μόνο μια γενική δήλωση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα των δημιουργών αλλά και των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων. Επομένως, ε, θα ψηφίσω το κείμενο, ε, γιατί παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προστατεύσουν τα δικαιώματα των δημιουργών, αν και θα ήθελα και κάτι παραπάνω για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση εδώ ε, δείχνει πόσο πάθος ε, μας χαρακτηρίζει στον κοινοβουλευτικό μας βίο. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, ε, αλλά σίγουρα δεν βαρεθήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Τα δικαιώματα των πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να προσαρμοστούν στην σύγχρονη πραγματικότητα. Και υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν κερδίζουν πάρα πολλά, που δεν γράφουν το best seller και έχουν ε, Λογαριασμού ε, εκατομμυρίων. Για αυτούς ε, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επισφαλής και ιδίω ό,τι αφορά τα πνευματικά του δικαιώματα. Εμείς θέλουμε όχι να καταστρέψουμε το ελεύθερο διδίκτυο, αλλά να προστατεύσουμε τα δικαιώματα. Θέλουμε επίσης όλοι να, να προστατεύσουμε την ελευθερία έκφρασης για όλους, αλλά θέλουμε ε, και την προστασία των δημιουργών. Θέλουμε ευθύνη για τις ε, πλατφόρμες. Αυτό οδηγεί όμως σε φιλτραρίσματα, ε, στο upload filters. Εγώ θεωρώ ότι σε όλο αυτό είναι η σημασία η κεντρική που έπρεπε να έχει προστασία των δημιουργών. Άρα πρέπει να υπάρχει δίκαιη αναλογική αμοιβή για τους δημιουργούς. Γι' αυτό δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα της προφορίας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Μπαίνουμε στη διαδικασία. Ε, catch Η πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Σόιντρόβα. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Άξελ Φως, τον εισηγητή για την ευσυνείδητη εργασία του και το γεγονός ότι ήταν πολύ θαραλέος γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη εκστρατεία. Ε, Πιστεύω λοιπόν ότι έχει φτάσει σε μια εξισορρόπηση μεταξύ πλατφορμών, δημιουργών και ημών των χρηστών. Οι μη εμπορικές πλατφόρμες όπως ο Wikipedia και άλλες έχουν γίνει αποδεκτές και το άρθρο 13 τάσεται κατά της λογοκρισίας. Αυτοί που αντιτίθενται δεν προβάλλουν μία ε, επιχειρηματολογία. Πώς όμως θα αμείβονται σωστά οι δημιουργοί αν δεν υπάρχει το άρθρο 13. Εμείς θα πρέπει να έχουμε πολύ ε, καλής ποιότητας ε, έργαση. Η κυρία Κονέτσνα προβάλλει μία μπλε κάρτα και δεν προβλέπεται στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Σόιντροβα την δέχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σόιντροβα αν μιλά για μια συντονισμένη καμπάνια τι εννοεί όταν μιλά για εκδότες, εκδότες που απειλούν τους δημοσιογράφους και στην περίπτωση αυτή θα υπάρξουν συνέπειες, δηλαδή αν υπάρχει έλεγχος περιεχομένου. Τι εννοείται, πρόκειται για μία ποταπή συναλλαγή, τίποτα άλλο. Απλώς έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Κυρία Σόιντροβα, θα ήθελα να πω ότι ότι ε, εκτιμώ σε αυτή τη συζήτηση τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το ανοιχτό πνεύμα και τη διάβια. Αν εσάς μπορούν να σας εκβιάσουν, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εγώ δεν υφίσταται κανέναν εκβιασμό. Πρέπει να βρούμε μια δίκαιη λύση για όλους τους δημιουργούς. Δεν θα πρέπει να δεχθούν δεχόμαστε κακόβουλους χειρισμούς. γκιλάρια ένα λεπτό μετά από ε, τρία χρόνια εργασίας θα πρέπει να φτάσουμε σε μια λύση που να είναι δίκαιη και εξισορροπημένη. Αλλά δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα όμως και η ελευθερία του εκφράζεστε, η καλλιτεχνική δημιουργία, το έρευνα. Αυτό λέει το Σύνταγμά μας, αλλά και η Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και φυσικά η αλυσίδα αξιών είναι η δημιουργή έναντι των γιγάντων του διαδικτύου που χρησιμοποιούν τα δεδομένα και δεν καταβάλουν φόρους, χρησιμοποιούν τρόλ έτσι ώστε να εξοριγνύουν στοιχεία. Μετά από αυτή την οδηγία, θα υπάρχει όμως το διαδίκτυο, αλλά και η ελευθερία του εκφράζεστε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνιο Ιππίντο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, εγώ κατανοώ τη θέση των Γάφα, Google, ε, Apple, Facebook και Amazon που όλοι αντιτίθενται σε αυτή την οδηγία γιατί απειλεί τα δυσθεώρητα κέρδη στα οποία έχουν φτάσει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή προστατεύεται το περιεχόμενο των δημιουργών, εκδοτών και συγγραφέων. Καταλαβαίνω γιατί η γκάφα αντιτίθενται σε αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κόμματα πειρατών, κόμματα κατά της δημιουργίας και των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Και καταλαβαίνω γιατί και η άκρα δεξιά αντιτίθενται σε αυτά τα ε, πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την, τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Καταλαβαίνω γιατί η άκρα δεξιά αντιτίθεται. Πιμέντο Λόπες. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα συμφέροντα των γιγαντιαίων οργανισμών όπως, όπως η Google και η Amazon που δεν δέχονται τη σωστή αμοιβή των δημιουργών. Πρόκειται για ε, επισφαλή εργασία πλέον των δημιουργών και ε, δίδεται ένα θεσμικό πλαίσιο σε αυτά τα φίλτρα, ενώ υπάρχει συγκέντρωση και μονοπόλιο του ψηφιακού τομέα. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε τους δημιουργούς, τους εκδότες, τους συγγραφείς και ούτω καθεξής, για να μπορούν να αμείβονται σωστά μέσα στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού του πολιτισμού με τη διάδοση περιεχομένου χωρίς ε, φίλτρα και λογοκρισία που ε, προωθούν οι μεγάλες πλατφόρμες που φημώνουν τους δημιουργούς. Η κυρία Βερκούνεν για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η οδηγία δεν είναι τέλεια. Είναι από το κόμμος πέντε ετών διαπραγματεύσεων και συμβασμών. Ευχαριστώ θερμά τον Άξελ για το έργο του εν μέσω αντιπαρατηθημένων απόψεων. Θεωρώ ότι προστατεύει παρκώς τα δικαιώματα των δημιουργών ε, Πρόεδρος, ξεκινήστε παρακαλώ από την αρχή λόγω τεχνικού προβλήματος. Κυρία Πρόεδρε, έλεγα ότι η οδηγία δεν είναι τέλεια. Σπάνια έχουμε να κάνουμε τέλεια νομοθετήματα. Είναι από το κόμμα 5 των διπλωματεύσεων. Συγχαίρω και ευχαριστώ τον Άξελ Φως και όλους όσους συνέβαλαν στο έργο αυτό. Πετύχαμε πολλά. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημιουργών και στην ψηφιακή εποχή. Αυτή είναι μια καλή αρχή. Και επίσης να θυμίσω ότι η οδηγία δεν θίγει την ελευθερία της έκφρασης. Δεν θέτουμε τροχοπέδι σε τίποτα. Έχουμε πλατφόρμες βεβαίω, εμπορικές. Εκεί βάζουμε όρια. Και αυτό είναι καλό και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Κέπχαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγοι για τους οποίους ε, δεν πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτή την οδηγία. Οι νοφείς επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν εξαιρούνται και μετά από τρία χρόνια θα πρέπει ε, να αναλάβουν και να καταστήσουν αυτά τα φίλτρα των μεγάλων επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλο επιχειρηματικό ε, μοντέλο, πολύ επιτυχημένο για τους Αμερικανικούς κολοσσούς. Δεν το θέλουμε όμως, αλλά δεν είμαστε υπέρ της οδηγίας και για κάτι ακόμη, γιατί τελικά δεν φαίνεται να έχει ως στόχο την αναλογική αμοιβή των καλλιτεχνών και δημιουργών. Τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία σε αισθητολογικέ σκέψει έχουν εντελώ αποδυναμωθεί ω προ την ισχύουσα διατύπωση. Αντίθετα, εμεί θέλουμε ισχυρότερα δικαιώματα για του δημιουργού. Αυτά δεν εξασφαλίζονται όμω, αλλά μόνο όσοι εργάζονται ε, σε εκδότε ε, είναι ε, αντικείμενο προστασία και οι επόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίε δηλαδή δεν έχουν αυτή την προστασία και αυτό είναι λάθο. Και κυρία Κώστα, τελευταία ομιλήτρια στο ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ευχαριστώ. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, να κατανοήσει ο κόσμος ότι οι δημιουργοί ε, με τη σειρά τους δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται και να υποαμείβουν την εργασία των άλλων. Δεν έχει νόημα να υπάρχει εκφοβισμός κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρουμε ότι σήμερα θέλουν να υπερασπιστούν τα εμπορικά τους δικαιώματα. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη πλατφόρμα έχει ε, υπέρογκα έσοδα από τη διαφήμιση αλλά η Silicon Valley δυστυχώς όπου και αν βρίσκεται ανά τον κόσμο δεν καταβάλει φόρους. Δεν ήθελα να σας σταματήσω, απλώς να επιβραδύνετε λιγάκι. Έχετε 15 δεύτερα στη διάθεσή σας, αλλά μιλάτε με ταχύτητα φωτός, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα 15 δεύτερα. Δεν σας ακούω, κυρία Κώστα. Έχετε 15 ε, δεύτερα. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι πρόβλημα για μένα. Για μας πρόκειται για μια μεγάλη μάχη για την δημιουργία και τον πλουραλισμό της πληροφορίας. Υπερασπιζόμαστε εκατομμύρια θέσεων εργασίας ε, για τους εκδότες, ε, δημιουργός και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε καταστήλει πολλά fake news, ε, τα οποία θα πρέπει να κατασταλούν. Η Wikipedia πολλές φορές παραπλανά. Κύριε Φρίερ, Υπάρχει μια σύγχυση εδώ γιατί δεν σας είχα στον κατάλογο μου. Θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Ward, υπάρχουν τόσοι άλλοι που δεν μπορεί να γίνει. Ας ελέγξουμε τις υπηρεσίες πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί ξέρω ότι το θέμα είναι σημαντικό για τους συναδέλφους. Παρακαλώ, κύριε. Ένα λεπτό αυστηρά. Θα πρέπει να θυμηθούμε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η οδηγία. Όχι γιατί υπάρχει δυσκολία πρόσβαση στο ίντερνετ, αλλά επειδή οι πολίτες θέλουν να καρποθούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχει μεγάλη πειρατεία. Αυτό είναι έγκλημα γιατί δεν υπερασπιζόμαστε τους ε, κανόνες της παραγωγής ε, στην τέχνη, πολιτισμό και δημοσιογραφία αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όταν χρησιμοποιούμε μια εικόνα ή ε, ένα συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμά του. Εάν ο δημιουργός θέλει να υπερασπιστεί το έργα του, δεν έχει επαρκή μέσα για να το κάνει στον ψηφιακό χώρο. Είναι όνειδος αυτό, το ότι δεν δίνουμε τη δυνατότητα αυτή στους δημιουργούς. Γραπίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Καθίσταται σαφές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέα τον οποίο θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Όλα ξεκίνησαν από την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία του εκφράζεστε, αλλά και προστασία του δημιουργού και ανταμοιβή της εργασίας. Χρειαζόμαστε όμως και μία δημιουργική βιομηχανία. Δεν μπορούμε χωρίς πολιτισμό. Βεβαίως, τα άρθρα 11, 13 και 14 είναι χρήσιμα. Όλοι συζητήσαμε με όλους και θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτά τα άρθρα για να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και να βελτιώσουμε αυτή την οδηγία. Αν δεν κάνουμε όμως τίποτα, δεν νομίζω ότι η ψηφική αγορά θα προστατευτεί περισσότερο. Δεν θα ε, προστατεύσουμε τους δημιουργούς. Τα άρθρα αυτά έχουν αλλάξει καπούτο ένα λεπτά. Ξέρω ότι μερικοί είναι δυσαρεστημένοι που δεν θα τους δώσω το λόγο. Καπούτο. Είναι τρίτη φορά που παρεμβαίνω για την οδηγία copyright. Στην αρχή μίλησα για αναπομπή στην Επιτροπή για καλύτερη εξισορρόπηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση αναπαραγωγής. Η οδηγία για την πνευματική οδιοκτησία θα βοηθήσει στην ανταμοιβή των δημιουργών. Αυτή τη στιγμή δέχομαι χιλιάδες mail από διάφορα λόμπι για να ε, συνεχίσουν τα προνόμια που είχαν κατά το, τα πρώτα χρόνια του 2000, την πρώτη δεκαετία δηλαδή. Ε, και γι' αυτό δεν νομίζω ο, παρά να λάβουμε υπόψη τους τριμερείς όπου απαγορεύεται η λογοκρισία και υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο διαδίκτυο και για όλες τις πλατφόρμες. Η κυρία Γκουιλάρ Γκαρθία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συζήτηση και αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ ε, αμφιλεγόμενη και επίμαχη. Όχι γιατί υπάρχει απόκληση απόψεων, κάτι που είναι καλό σε κάθε συζήτηση, ήθιστε να υπάρχουν αποκλήσει απόψεων, αλλά είναι πολύ περίεργο. Μιλάμε για έναν απαραίτητο κανονισμό που θα ρυθμίσει την ψηφιακή αγορά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο πάθος. Εμένα κάπως με ξενίζει, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στρέβλωση στην ενιαία ψηφιακή αγορά και με τον κανονισμό, με την οδηγία μάλλον αυτή, στόχος είναι ε, προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και νομίζω ότι είναι ισορροπημένη πρόταση. Γιατί είμαστε λοιπόν αντίθετοι σε αυτή τη ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν σημαίνει απαγόρευση, Απλά σημαίνει ότι μπαίνουν κανόνες, έτσι ώστε όλοι σε αυτήν την αγορά και στη ψηφιακή αγορά ε, και στην εμπορική και τη χρηματοπιστωτική αγορά να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μόνο περί αυτού πρόκειται. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ ε, της οδηγίας αυτής. Ευχαριστώ κυρία Ward. Ως εκπρόσωπος των εργατικών για τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι πρέπει να υπερμηνθούμε των μικρομεσαίων που εργάζονται στο δημιουργικό. Πρόκειται εδώ για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση εδώ και 15 χρόνια και θα σταματήσει επίση του γίγαντε από τι επεμβάσεις του στο διαδίκτυο. Ακόμη πιο σημαντικό, διασφαλίζει η οδηγία, ότι οι δημιουργοί απολάβουν αξιοπρεπού αμοιβή. Αυτό το πακέτο μεταρρύθμιση κάνει κάτι επιτέλου για την σημερινή κατάσταση όπου ένα τραγούδι μπορεί να, να μεταδοθεί 5 εκατομμύρια φορές πριν ο δημιουργός του μπορέσει να διεκδικήσει κάποια αμοιβή. Αυτό θέλουμε, να αναγνωριστούν και να μειωθούν επαρκώς οι δημιουργοί. Η, η οδηγία αυτό κάνει, αποτελεί επένδυση στην, στον τομέα του δημιουργικού. Θέλω να ευχαριστήσω τις ενώσεις των καλλιτεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο Διακόπτη πρόεδρος. Πρέπει να σας διακόψω και τώρα ο Επίτροπος Ανσίπ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συζήτηση. Πολλοί μιλητές αναφέρθηκαν στο φίλτρο, στο περίφημο φίλτρο το οποίο δεν αναφέρεται όμως στο κείμενο της οδηγίας. Όπως γνωρίζουμε, χρησιμοποιείται από τις μεγάλες πλατφόρμες η καταψήφιση της οδηγίας δεν θα καταργήσει τα φίλτρα αυτά. Η οδηγία των αντίων θα δώσει στους πολίτες μας το δικαίωμα να ζητήσουν την αφαίρεση υλικού για το οποίο πρέπει να λάβουν αμοιβή. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Η ψηφοφορία αφορά το μήνυμα που θέλει να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δημιουργούς της. Και είναι απλά τα πράγματα. Φροντίζουμε για εσά, σας έχουμε στο μυαλό μας και σας προστατεύουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε το πολύτιμο έργο σα και να συμβάλλετε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι θεμέλιο της κοινωνίας μας. Είναι πηγή των αξιών μας και της έμπνευσή μας. Η τελική δικαιούχη, αν θέλετε, αυτής της οδηγίας είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σύγχρονο περιβάλλον για τα πνευματικά δικαιώματα σημαίνει πρόσβαση στην ψυχαγωγία, στην δημοσιογραφία και Γι' αυτό το λόγο η ψηφοφορία αφορά τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει τις πολύπλοκες νομικές προκλήσεις του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις και αυτό είναι καλοδεχούμενο στο πλαίσιο ενός διαλόγου. Αφού γραστήκαμε τις διστάμενες απόψεις, δείχνουμε σεβασμό όμως πιστεύουμε ότι εν τέλει το κείμενο από το του τριμερούς διαλόγου είναι ισόρροπο και επιτελεί ακριβώς τον στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή, τον εξυγχρονισμό του δικαίου μας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να ετοιμαστούμε για την ψηφιακή εποχή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους και οδησίες ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Άνσιπ. Καλωσορίζω όλους και πάλι. Συνέχιζω να προεδρεύω κύριος Φως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στη σημερινή συζήτηση ε, και από κάποιες παρεμβάσεις ε, ξαναβλέπουμε ότι κάπως έχασε το μέτρο αυτή η συζήτηση. Δεν θα υπάρξει λογοκρισία με αυτή τη μεταρρύθμιση η ε, ελευθερία έκφραση, η νόμιμη, δεν θα περιοριστεί με αυτή την έκθεση. Εμείς καταφέρνουμε να έχουμε ε, ασφάλεια δικαίου ε, και νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, οι χρήστες, οι πολίτες έχουν περισσότερα δικαιώματα και ελευθερία, Facebook, Google, YouTube κτλ. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν παραπληροφορούν και βάζουν πάρα πολλά λεφτά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και δείχνουν πόσο εύκολο τελικά είναι τις ε, ε, ομάδες των νέων, την νεολαία να τις ε, χειραγωγήσουν και ε, να τις επηρεάσουν. Σήμερα ε, το Κοινοβούλιο, η Δημοκρατία μας ε, δεν στρέφεται κατά τον, και δεν θέλει να επιβληθεί σε βάρος των κολοσσών του διαδικτύου, αλλά να εξασφαλίσει την προστασία της πνευματικής δεξίας. γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την πνευματική δεξία, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θέλουμε δίκαιη αμοιβή των δημιουργών. Αυτή είναι η στόχη μας και είναι στο δικό μας χέρι σήμερα να σώσουμε ε, την ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία. Δεν θέλουμε εκμετάλλευση από τα μονοπόλια. Ε, στο χέρι μας είναι σήμερα να προσφέρουμε την ε, απαραίτητη και την αναγκαία προστασία στους κλάδους της δημιουργικής πολιτιστικής βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Φως, λέει ο πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε